il presidente η συνεδρία σας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διερεμηθεί. Παρατηρήσεις υπάρχουν. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή επί τη ευκαιρία τη παρουσίαση του προγράμματο δραστηριοτήτων τη Προεδρία τη Ρουμανία. Και επί τη ευκαιρία θέλω να καλωσορίσω την Πρωθυπουργό τη Ρουμανική ε, Δημοκρατία, την παλαιά συνάδελφο κυρία Νταντσίλα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας ως Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Ανέλαβα την εντολή της Προεδρίας από την Αυστρία και θα ήθελα να πω με αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ μάλλον στις ευχαριστίες μου προς την Αυστριακή Προεδρία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Φιλανδία και την Κροατία γιατί είχαμε μία πολύ καλή συντονιστική δραστηριότητα για ένα κοινό πρόγραμμα για τους ε, επόμενους 18 μήνες. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη ήξερε από πάντα να ξεπεράσει προς κόμματα και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βασίστηκε στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Σήμερα βρισκόμαστε εκ νέου στη πολλωστή διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Όπως ξέρετε, κάθε τέτοια κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και νέα αρχή. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω ότι ότι σύμφωνα με το δικό μας όραμα για τους επόμενους έξι μήνες ε, δεν ε, μιλάμε απλούστατα για μία επίσημη εντολή. Έχουμε 500 εκατομμύρια που αναμένουν απάντηση από την Ευρώπη. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εργάζονται για τους πολίτες και φτάνουν σε αποτελέσματα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Γνωρίζω ότι το πρώτο στάδιο της εκπεριτροπής προεδρίας θα, είναι, θα αποτελείται από εντατική εργασία σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό βασίζουμε στη δική σας υποστήριξη για να ολοκληρώσουμε πολλά θέματα που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε προκλήσεις. Το δικό μας πρόγραμμα βασίζεται στην συνοχή ως κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις, διαστάσεις πολιτική, έτσι ώστε να υπάρχει ένωση μεταξύ κρατών μελών, οικονομική και εδαφική συνοχή και μείωση των πολλαπλών ταχυτήτων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών καθώς και κοινωνική συνοχή για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις τέσσερις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η πρόσληψη πραγμάτων θα πρέπει να ακολουθήσει μία εγκάρσια πορεία με βάση τις θεματικές μας και με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες, δηλαδή Ευρώπη της σύγκλησης, της ασφάλειας, της Ευρώπης των κοινών αξιών και του παγκόσμιου παράγοντα. Η Ευρώπη της σύγκλησης είναι ο πρώτος πυλώνας δράσης της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο για την διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανέλυξης και μείωση ανισοτήτων, ανταγωνιστικότητα και συνδεσιμότητα καθώς και ένωση των αγορών. Αυτό είναι ο πυρήνας της, οικονομικής, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ένας από τους στόχους της Ρουμανικής Προεδρίας είναι να προωθήσει τα νομοθετικά ζητήματα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς για να έχουμε μία χρηστή λειτουργία της αγοράς. Θα πρέπει να παγιοποιήσουμε την επιστημονική και τεχνολογική βάση των βιομηχανιών έτσι ώστε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας. Αυτό αφορά και την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ψηφιακή επίθεση έχει προωθηθεί ήδη και από τους Εσθονούς και τους Αυστριακούς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπό τον ίδιο ρυθμό. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη λειτουργική διασύνδεση Ανατολής Δύσης, Βορρά και Νότου για να προωθήσουμε αυτές τις τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και προώθησης των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών. Θέλουμε μία νέα πολιτική στον βιομηχανικό τομέα, αλλά έχει μεγάλη σημασία και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς. Αυτά τα θέματα κατέχουν έχουν σημαντική θέση στην Προεδρία μας. Ο δεύτερος πυλώνας της Ρουμανικής Προεδρίας αφορά την Ευρώπη της ασφάλειας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που απειλούν τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και απειλών που υποσκάπτουν την ευημερία της ανοιχτής μας κοινωνίας. Σε έναν κόσμο σε ψηφιοποίηση θα πρέπει να προωθήσουμε την προστασία των πολιτών στον εικονικό κόσμο. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε την ανθεκτικότητα της Ένωσης ως προς τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία για οποιοδήποτε πρόγραμμα που αφορά τον τομέα της ε, πληροφορικής. Στο πλαίσιο της ασφάλειας θα προωθήσουμε και τις διαπραγματεύσεις μας και τις πρωτοβουλίες για να έχουμε μία συνεκτική προσέγγιση των ορών της ε, μετανάστευσης, την ενδυνάμωση των συνόρων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση της ασφάλειας των πολιτών στον εικονικό κόσμο, καθώς και επέκταση της εντολής της Ευρωπαϊκής εισαγγελία σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επίσης, συνεργασία της δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστικών αρχών στο θέμα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Θα θέλαμε λοιπόν να προωθήσουμε τη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες ε, διαμετακόμισης στα πλαίσια των μεταναστευτικών ρών. Το τρίτο θέμα είναι η Ευρώπη ως παγκόσμιος ε, δράστης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινέ ε, αποφάσεις όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας θα θέλαμε να ενισχύσουμε την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια ενός συμπληρωματικού χαρακτήρα δράσης ως προς το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχέσεις άμεσης γειτονίας για να προωθήσουμε τις δράσεις μας. Δέκα χρόνια μετά τις εταιρικές, δέκα χρόνια μετά την απαρχή των εταιρικών σχέσεων με τις ανατολικές χώρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια. να δούμε και ποια θα είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκακέρα. Να συγχρονίσουμε το πολυμερές εμπορικό πλαίσιο καθώς και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο. Μιλάμε για μια Ευρώπη κοινών αξιών. Για να προωθήσουμε λοιπόν την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίσει η κοινωνία μας όπως ο ε, ρατσισμός, μυσαλλοδοξία, ξενοφοβία, αντισημιτισμός και ρητορική μίσους θέλουμε μία πιο δημοκρατική κοινωνία, γι' αυτό θα μιλήσουμε για ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων, όπως επιθυμούν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για την αξιοπιστία μας εναντί των πολιτών. Αυτό το λέω και από την πλευρά της Ρουμανίας, την οποία εκπροσωπώ και ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει μια άνηση μεταχείριση της ε, Ρουμανίας τη στιγμή που επικρίνεται η χώρα μας για θέματα τα οποία γίνονται ανεκτά όσον αφορά άλλα κράτη-μέλη και για τη Ρουμανία υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ρήτρες αιρεσιμότητας που δεν ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης παραμένουμε εκτός χώρου Σέγγεν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ζαν Κλόντ Γιούνκερ και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη γιατί μας υποστήριξαν για την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Αυτά όλα τα αναφέρω για να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες ευρωπαϊκές αποφάσεις συρρυκνώνουν το πλαίσιο δράσης συγκεκριμένων πολιτών και μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους πολίτες των κρατών μελών που εμπλέκονται και δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση πολιτών κρατών μελών. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν το κλειδί δράσης μας σε ατομικό επίπεδο και συλλογικό μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινή μας δραστηριότητας. Θα πρέπει οι νέοι να συμμετέχουν στη διαδικασία οικοδόμησης μιας δυνατής Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι παρακολουθούμε τις αποφάσεις ε, του Βρετανικού Κοινοβουλίου ως προς το Brexit και είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει άμεσα τη Ρουμανική Προεδρία. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη τα νέα αυτά δεδομένα και θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κατάσταση. Το Μάιο Επίσης θα εκλεγεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη αυτή τη νέα εκλογική διαδικασία γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε μία πιο δυνατή Ευρώπη με βάση τις ιδρυτικές ε, αξίες της και με βάση τις ευρωπαϊκές γενικότερα αξίες. Πιστεύω σε μια Ευρώπη μέσω της ενότητας, μέσα στα πλαίσια της τήρησης των εντολών και καθηκόντων και πιστεύω σε μια πιο ευρωπαϊκή Ευρώπη μέσα στα πλαίσια των κοινών αξιών και τη συμμετοχής των πολιτών που θα πρέπει να νιώθουν ότι ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο μία ενωτική Ευρώπη, μία ενωμένη Ευρώπη στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα που αποτελεί μία πολύ καλύτερη λύση για όλα τα μελλοντικά μας προβλήματα και την αντιμετώπιση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. La λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας εκ μέρους του Πρόεδρου Γιουνκέρ, εκφράζω την χαρά και ικανοποίησή μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την πρώτη στην ιστορία Ρουμανική Προεδρία. Η Ρουμανία, όπως και η Εστονία, η πατρίδα μου, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, γιόρτασαν την εκατοστή του επέτειο πέρσι επέτειο από την ίδρυση. Στιγμή σημαντική για να κοιτάξουμε και προς, το, προς τα πίσω, να δούμε τι έδαφος έχουμε διανύμησει σε αυτά τα χρόνια. Η Ρουμανία έχει διανύσει σημαντικό έδαφος λοιπόν και βρίσκεται τώρα στη θέση που της ανήκει, στο κέντρο της Ευρώπης. Καλύτερο σύμβολο αυτής της προόδου δεν μπορούσε να είναι άλλο από την Προεδρία αυτή στο επόμενο εξάμεινο η Ρουμανία θα ηγηθεί του Συμβουλίου των Υπουργών σε μια κέρια σημασία εποχή για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι με τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπή στο σύνολό τη, όπου παρακολουθήσαμε και το πολύ καλό επίπεδο των προετοιμασιών, αλλά και τον ενθουσιασμό που εμπνέει την κυβέρνηση για το έργο που έχει μπροστά τη. Προεδρία όμως σημαίνει ταυτόχρονα και ευθύνε πάνω απ' όλα σε περίοδους ε, αλλαγών, εξελίξεων και προεκλογικών εκστρατιών. Όπως πολλές φορές έχει επισημάνει ο πρόεδρος Γιονκέρ, η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας. Είναι έτοιμη να σας στηρίξει σε κάθε βήμα της πορείας σας. Θα εργαστούμε χέρι με χέρι με όλα τα θεσμικά όργανα, με όλους τους θεσμούς και τις... Ε, τους αρμοδίους που θα εμπλακούν σε αυτήν την ε, Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Μπορείτε να υπολογίσετε λοιπόν σε εμά. Όπω όμω υπολογίζετε εσεί σε εμά, μπορούμε και εμεί να υπολογίζουμε σε εσά. Υπολογίζουμε στο ιδιωτικό σα πνεύμα, τη σταθερότητά σα, την ικανότητά σα να χτίσετε γέφυρε, να οικοδομήσετε συνένεση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στα εσωτερικά σα. Και αυτό το λέω γιατί κάθε επιτυχημένη Προεδρία πρωταρχικά και πάνω απ' όλα εξαρτάται από την εθνική ενότητα και την πολιτική συνένεση. Ένα ενωμένο μέτωπο λοιπόν στο εσωτερικό της χώρας θα βοηθήσει να προχωρήσει μια ενωμένη Ευρώπη. Η Ρουμανία γνωρίζει καλύτερα από πολλές άλλες χώρες το δύναμη της ενότητας. Κατά την προετοιμασία για την ένταξη στην Ένωση στάθηκε ολόκληρη η χώρα ενωμένη και εργάστηκε για να εξασφαλίσει πως θα εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια προσχώρησης. Η επιχείρηση αυτή, η προσπάθεια αυτή δεν ήταν απλώς μία ε, επιβεβαίωση σε κουτάκια των ε, προϋποθέσεων που πρέπει να πληρωθούν. Ήταν η προετοιμασία για ένταξη σε μια ένωση κοινών αξιών, ελευθερίας, δημοκρατίας, κράτους δικαίου, αυτών των αξιών για τις οποίες αγωνίστηκε η χώρα, αυτών των αξιών που ποτέ δεν μπορούν να ε, μειωθούν ή να αποδυναμωθούν. Το επόμενο εξάμεινο, αλλά και πέρα από αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Αξιότιμοι βουλευτές, άρχισα την ομιλία μου λέγοντας ότι κάθε Προεδρία συνοδεύεται από ευθύνη για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό θα είναι το καθήκον της Ρουμανίας στο επόμενο εξάμεινο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο στο μέλλον. 242 προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν κατατεθεί πρέπει να εγκριθούν από τους συνομοθέτες. Θα είναι πολύ περιορισμένο το διάστημα αυτό που θα έχετε στη θέση σας για να καλύψετε αυτά τα καθήκοντα καθώς το Κοινοβούλιο 18 Απριλίου σταματάει τις εργασίες του για να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Αυτές οι 242 ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγαλύτερο τους ε, τμήμα αφορούν πάρα πολύ σημαντικά κέρια για την Ευρώπη θέματα όπως ε, το Brexit, η μετανάστευση και άλλα. Ο δικό μου τομέα τη ψηφιακή οικονομία έχει περίπου 30 προτάσεις που πρέπει ακόμη να εγκριθούν. και αφορά πάνω απ' όλα προτάσεις που θα φέρουν σημαντικές αλλαγές, ουσιαστικέ αλλαγές στην καθημερινή ζωή του Ευρωπαίου. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει, κάνει κανείς αγορές πέραν των συνόρων ηλεκτρονικά το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικής ζωής στο διαδίκτυο, της προστασίας από τις κυβερνοεπιθέσεις, περιλαμβάνεται σε αυτές τις προτάσεις. Εταιρικοί κανόνες ε, που έχουν τα χαρακτηριστικά των κανόνων του 21ου αιώνα. Κανόνες για τον ψηφιακό κόσμο σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για το προσοχή προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ δεν μιλούμε για αριθμού ή για δεκαδικά ψηφία. Εδώ μιλούμε για αποφάσει που θα κρίνουν το μέλλον τη Ευρώπη, θα ορίσουν το τι είδου Ευρώπη θέλουμε για το μέλλον. Είναι το μέλλον μα, εκφρασμένο σε αριθμητικού όρου. Γιατί ο προπολογισμό θα δείξει στον Ευρωπαίο ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πάρει στα χέρια τη το μέλλον τη. Όταν ε, συνέλθουν στο Συμπίου στις 9 Μαΐου οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να είμαστε θέση να δείξουμε πως έχουμε προοπτική για μέλλον, για ένα μέλλον πιο ισχυρό, πιο ενωμένο, ένα, ένα μέλλον μιας Ευρώπης με ηγετική θέση και ενωμένη. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα πάρει μαζί του Ευρωπαίος όταν προσέλθει στην Κάλπη, λίγες μόνο εβδομάδες αργότερα ιδιαίτερα για αυτούς που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν, θα έχει κρίσιμη σημασία. Είτε πρόκειται για ψηφοφόρους του, των κρατών της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά ή του Νότου της Ευρώπης, όλοι αυτοί οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θέλουν ένα μέλλον πιο φωτεινό, πιο αισιόδοξο. Θέλουν μια Ευρώπη ενωμένη, που θα αναπνέει με τους δύο τις πνεύμονες, και τον Ανατολικό και το Δυτικό, που θα ενώνει όλες τις πλευρές της Ευρώπης. Πρέπει να τίνουμε λοιπόν χείρα βοηθεία σε αυτούς τους νέους, να τους δώσουμε το χέρι και να τους δείξουμε ότι η Ευρώπη αναπτύσσεται για το δικό τους καλό. Και αυτό είναι το καθήκον που έχει να επιτελέσει η τρέχουσα Προεδρία της Ρουμανίας. Γι' αυτό θέμαστε στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουμε να το υλοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μουτσομέσικα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Τόλογιαν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλωσορίσατε κυρία Πρωθυπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδροι των ε, θεσμικών οργάνων σας ε, υποστήριξαν, εξέφρασαν την υποστήριξή τους εκ των προτέρων της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Μετανάστευση, κινητοποίηση στις μεταφορές και περίπου 40 εκθέσεις που αφορούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 και από τις λύσεις που θα δοθούν, οι λύσεις μάλλον που θα δοθούν, θα αποτελέσουν πρόκριμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πορείας της. Έχετε πολλούς νέους υπουργούς που δεν έχουν πείρα στις διαπραγματεύσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσετε από αυτούς τους υπουργούς να βασίζονται στις ε, συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της μόνιμης ρουμανικής αντιπροσωπείας που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά. Μιλήσατε πολύ σωστά για την ανησυχία που υπάρχει ως προς τις πρώην ανατολικές χώρες που δεν θα πρέπει να μείνουν στο απόκεντρο της ένισης. Αλλά, όπως ξέρετε, η Ρουμανία δεν ανήκει ούτε στην Ευρωζώνη, ούτε στο χώρο Σέγγεν. Άρα είναι πλήρες μέλος, αλλά με σοβαρές ελλείψεις. Οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τόνισαν ότι θα υποστηρίξουν τη Ρουμανία στην προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Όμως, ως Πρωθυπουργό έχετε υποχρεώσεις έναντι όλων των πολιτών της Ρουμανίας και του επιχειρηματικού χώρου να συναντηθείτε με τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας και της Γαλλίας, με τους καγκελάριους της Αυστρίας και της Γερμανίας και να τους πείσετε ότι η Ρουμανία είναι έτοιμη να προσχωρήσει στο χώρο του Σέγγεν. Στην Ολλανδία θα πρέπει να μεταβείτε και στη Βουλή των Κοινοτήτων και επίσης δεν υπάρχει αξιοπιστία τη, όπως ξέρετε, του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα της Γερουσίας. Ως προς την Ευρωζώνη, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας προσχώρησης, είπατε ότι θα δημοσιοποιήσετε το πρόγραμμα δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2018 παρήλθε και δεν έχουμε ακόμα αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην άσκηση της Ρουμανικής Προεδρίας. Εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ούντο Μπούλμαν έχει το λόγο. Αγαπητή Πρωθυπουργέ, αγαπητή Βιορίκα, καλώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχαρητήρια επί τη ευκαιρία της ε, ανάληψης ε, της Προεδρίας από τη Ρουμανία. Όλοι γνωρίζουμε την προσωπική σας ε, αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρώην συνάδελφο σας γνωρίσαμε ως πάρα πολύ στρατευμένη Ευρωπαία και πραγματικά αυτό αποτελεί τη βάση για μια αγαστή συνεργασία μας με τη Ρουμανική Προεδρία δεδομένων και των όσων μας περιμένουν που τα αναφέρατε και της σοβαρή κατάσταση σε πολλούς τομείς πολιτικής. Άκουσα την ομιλία σας με ενδιαφέρον και έχετε δίκιο. Η περιφερειακή συνοχή, η κοινωνική συνοχή είναι ένα θέμα αποφασιστικό και εγκάρσιο. Και αυτή η ιδέα να οργανώσουμε με νέο τρόπο την ευρωπαϊκή σύγκληση θα πρέπει να κυριαρχεί στις συζητήσεις μας. Οι τελευταίες ώρες σήμερα έδειξαν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Λονδίνο και πόσο ακόμα έργο απομένει να γίνει μέχρι την ε, απόφαση απόψε. Θέματα φορολογικά, θέματα χρηματαγορών θα πρέπει να μας απασχολήσουν, να τα ε, επανακαθορίσουμε και το μεταναστευτικό είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Θα ήθελα εδώ να σας επενέσω και να αποτίσω ένα φόρο τιμής σας, γιατί κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αποφασίσατε να ενταχθείτε στο στρατόπεδο εκείνων που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στη Μεσόγειο, να σώζουν ζωές και όχι να εθελοτυφλούν απέναντι στα όσα συμβαίνουν ή να ενταχθούν στη λέσχη εκείνων που ήδη πανηγυρίζουν για την ε, διαφορία τους. Ε, θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε προβλήματα που έχουμε και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μας ανησυχούν. Πολλά ε, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Το δικαστικό σύστημα στη Ρουμανία θα πρέπει να παταχθεί, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά. Αν στην Ευρώπη υπάρχει τέτοια κατάσταση να επηρεάζουν οι μυστικές υπηρεσίες τη δικαιοσύνη και την εισαγγελία. Αυτό είναι απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι. Το αναφέρω εδώ, αλλά θα πρέπει να το συζητήσω και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, της Ρουμανίας, γιατί στη δική του αρμοδιότητα είναι μυστικές υπηρεσίες. Οπότε, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλή ε, ε, ομόνια, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και να αποδίνουμε και τις ευθύνες εκεί που ανήκουν. Τώρα θα μιλήσω για, ε, για πράγματα ε, τα οποία ορισμένοι λένε πίσω από την πλάτη κάποιον. Εγώ όμως τα λέω ξεκάθαρα εδώ. Αν στη χώρα σας υπάρχουν αδικίες από τη δικαιοσύνη, ε, θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι η απάντηση γενική αμνηστία, γιατί βάζει δίκιο και άδικο στο ίδιο τσουβάλι. Θα πρέπει να ε, κυριαρχήσει το κράτος δικαίου εκεί που χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Γνωρίζω ότι το επιθυμείτε και θέλω να σας ενθαρρύνω. Κάντε το αυτό γιατί ε, αυτό θα διευκολύνει και την Προεδρία σας και σας προσωπικά και τη χώρα σας και θα έχετε την Ευρώπη στο πλευρό σας αν το κάνετε. Το κράτος δικαίου είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών που προστατεύει τους ανθρώπους, εγγυάται τις ελευθερίες απέναντι στο κράτος και τερματίζει την αυθαίρετη κυριαρχία. Αυτό ισχύει έναντι όλων. Τα γνωρίζουμε εμείς αυτά οι σοσιαλδημοκράτες, γιατί 150 χρόνια αυτό ε, υπερασπιζόμαστε παντού όπου κινδυνεύει. Αλλά ε, το κράτος δικαίου ε, δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόφαση και πρόσχημα από τους πολιτικούς αντιπάλους για να γίνουν κάποια πολιτικά παιχνίδια. Κυρία Πρωθυπουργέ, εσείς είστε μια γυναίκα θαραλέα και το γνωρίζω. Η μεταρρύθμισή σας μπορεί να αποτελέσει θαυμάσια προϋπόθεση για τη συνεργασία μας στο επόμενο εξάμεινο. Και να πω κάτι σε κάποιους παντογνώστες εδώ, ιδιαίτερα ε, τους ανταγωνιστές σας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αν αυτές τις μέρες υπάρχει μια χώρα που κλείνουν πάλι πανεπιστήμια, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ από το φασισμό, ε, ε, που υπονομεύονται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, ε, και ε, φημώνεται ο κόσμος, τότε να πάτε να τα πείτε και στον κύριο Όρμπαν, γιατί δεν τολμάτε να το τα πείτε κατάμουτρα. Δεν χρειάζεται να σκουπίζετε τα παπούτσια σας στην ε, επερχόμενη Προεδρία. Είναι λάθος αυτή η κατάσταση. Η Ουγγαρία είναι το πρόβλημα. Τα είχα πει και στον κύριο Γιούγκερ προσωπικά. Έτσι θέλω να τα λέμε και αυτά εδώ. Εκ μέρου των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, κυρία Στίφενς. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρωθυπουργέ, καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά και να καλωσορίσω και τη Ρουμανική Προεδρία. Έξι μήνε είναι μια σύντομη περίοδο για να συζητήσει κανεί και να διαπραγματευτεί. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να συντονιστούμε μαζί με τι δύο επόμενε Προεδρίες. Για τη Ρουμανική Προεδρία η ευρωπαϊκή διεύρυνση είναι ήδη μια προτεραιότητα. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2018 εκφράζει την φιλοδοξία να διευρυνθεί. Αν κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, μπορούν έξι χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια να έχουν ενταχθεί περί το 2025. Καλύτερα όμως θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει κατά, ε, τάξη ε, στα εσωτερικά της. Και σας παραπέμπω στο Brexit που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών ε, για το μεταναστευτικό και την πολιτική μας. Για μας αυτή είναι η προτεραιότητα, η λάθρομετανάστευση. Και ε, παρακαλώ να ακολουθήσουμε το αυστραλιανό μοντέλο ε, που αποθαρρύνει τις παράνομες αφήξεις. Ελπίζω να συμφωνήσετε και να το συζητήσετε αυτό στις διαπραγματεύσεις ε, όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί το κοινοτικό κεκτημένο για το άσυλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Αλδέ ο Φερχόφστατ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ η χώρα σας αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια θα έλεγα πολύ κρίσιμη στιγμή αμέσως πριν τις ευρωεκλογέ. Έχω ετοιμάσει ένα κατάλογο πακέτο κινητικότητας και μεταφορών, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που χρειάζεται συμφωνία και βεβαίως πολύ σημαντικό δύο διαδικασίες άρθρο 7 μία κατά της κυβέρνησης της ε, Πολωνίας και μία που έχει ε, θέσει σε κίνηση το Κοινοβούλιο κατά της κυβέρνησης Ορμπάν. Πολύ δουλειά λοιπόν έχετε μπροστά σας και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί, να έχουμε και τρίτη περίπτωση άρθρου 7 κατά της Ρουμανικής κυβέρνησης αυτή τη φορά. Γιατί θα σας το πω. Έχω την εντύπωση πως δεν απέχετε πολύ από αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή καθώς συνεχίζετε να αγνοείται τις ε, γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας και ορισμένο για ορισμένα νομοθετικά ε, κείμενα, νομοθετικές προτάσεις που έχει ενώπιόν το ε, Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο της Βουλής και επικεφαλής του κόμματος, τον κύριο Τρεκνέ, ο ε, της τάσης της πλειοψηφίας σας είπε «Α, το κράτος δικαίου είναι θέμα ε, επικουρικότητας». Όχι, ένα λεπτό. Επικουρικότητα μπορεί να είναι για πολλά θέματα ισχυρός κανόνας, αλλά όχι για το κράτος δικαίου. Δεν εμπίπτει στην επικουρικότητα το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς το ίδιο, την ίδια ακριβώς μέρα, είπα και στον κύριο Ντερετσάνου, ο οποίος μου έδωσε την υπόσχεση πως η κυβέρνησή σας και τα δύο κόμματα που σχηματίζουν την κυβέρνηση συνασπισμού θα δεχθούν τις προτάσεις αυτές και θα συμμορφωθούν απολύτως στις νομοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πολλό συμφώνησε μαζί μου πως η Επιτροπή της Βενετίας θα κληθεί να ε, εκφέρει δεύτερη γνώμη άπαξ δηλαδή και οι προτάσει αυτέ προσαρμοστούν, θα αποσταλούν και πάλι στην Επιτροπή τη Βενετία. Και πρόκειται για προτάσει για την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, για τον ποινικό κώδικα, για την ε, ποινική δικονομία και για την νομοθεσία τη σχετική με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Θα πρέπει να σας επισημανώ με απόλυτη ειλικρίνεια πως από την ε, συνάντησή μας εκείνη που ήταν και ο κύριο Μπούλμαν και άλλοι στο, Βουκαρέ, καμία από τις ε, υποσχέσεις αυτές είναι δεμένα, υλοποιούνται. Η χώρα, η κυβέρνηση σας συνεχίζει στο δρόμο των χείριστων πρακτικών των άλλων, όπως του Ορμπάν και του Κασίνσκι. Και επιπλέον, σας ερωτώ, αληθεύει αυτό που διαβάζω στον τύπο, ότι δηλαδή σκοπεύετε να υιοθετήσετε νόμο που θα, χορηγήσει, θα χορηγεί αμνηστία για τις περιπτώσεις διαφθοράς δηλαδή οι μεγαλοκαρχαριές θα είναι εκτός του ελέγχου των δικαστηρίων. Ένα πολύ απλό πράγμα θα σας πω με την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η δική μου η πολιτική ομάδα και η πολιτική οικογένεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει το δρόμο της ε, συνένεση και δεν θα σας αφήσει ήσυχο. Θα θέλουμε να σταματήσει αυτή η πορεία. Θέλουμε να καθαρίσει η χώρα από τη διαφθορά και την κατάχρηση της εξουσίας από την παλαιά μυστική υπηρεσία. Και αυτό δεν αποτελεί επίκριση για τη χώρα ή το Ρουμάνο πολίτη, τους Ρουμάνους πολίτες. Είναι επίκριση κατά κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών της πολιτικής πλειοψηφίας που εκπροσωπείτε εσείς αυτή τη στιγμή. Και έχω κάθε δικαίωμα να το πράξω αυτό, να επικρίνω αυτές τις πρακτικές, γιατί είμαι επίτιμος πολίτης της Ρουμανικής Δημοκρατίας. Το 2001 μου ε, απονεμήθηκε, ύστερα από, την, ε, από τον αγώνα στον οποίο αποδίθηκα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί κανείς δεν μου το είχε ζητήσει, να προ, προσπιστώ τα δικαιώματα της Ρουμανίας μέσα από τη συνθήκη της νίκαιας, γιατί κάποιοι είχαν ε, την υπέροχη ιδέα, επειδή η Ρουμανία είναι χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, να τις περιορίσουν τα δικαιώματα, τις ε, ψήφους που τις αντιστοιχούν και μου χορηγήθηκε η ε, ιδιότητα του πολίτη, του επιτιμού πολίτη. Γιατί μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τα ε, ίδια δικαιώματα, ισότιμα δικαιώματα λοιπόν, για το, Ρωμένο, για το Ρωμανό πολίτη. Με την προσχώρηση. Μην το δείτε λοιπόν σαν επίκριση. Ακούστε αυτό που σας λέω και ακολουθήστε αυτούς τους αγώνες. Καταστείτε γνήσια πρωθυπουργός της χώρας σας. Καθαρίστε την ε, διαφθορά και την ε, βρώμα του παρελθόντος και έρθείτε σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της διαφθοράς. Ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων, η κυρία Σκακέλερ. Καλώ ορίσατε κυρία Πρωθυπουργέ και η Ρουμανική Προεδρία. Καλώ να ορίσει. Πάντα είναι μια ευκαιρία να λάμψει μια χώρα η Προεδρία και να δείξει ε, στις ικανότητές στη διπλωματία, στους συμβιβασμούς, στις προόδους και να εντυπωσιάσετε και με τις δεξιότητές σας ως χώρα και ως Πρωθυπουργός. Αυτό ε, είναι και βασικός μας ρόλος στις ε, θεσμικές σχέσεις και για να προχωρήσει η Ευρώπη. Αλλά η Προεδρία φέρνει και μια κυβέρνηση και μια χώρα στο προσκήνιο. Και αυτά που ανακαλύπτουμε για την ρουμανική κυβέρνηση μας ε, προκαλούν ανησυχία. Έχει μακρά παράδοση η Ρουμανία στον αγώνα για την ελευθερία και τις δημόσιες ελευθερίες. Απέταξαν μετά από 42 χρόνια μια δικτατορία οι Ρουμάνοι και η Ρουμανία έχει κάνει πολύ μεγάλες προόδους ε, κατά της διαφθοράς. Και μάλιστα οι Ρουμάνοι μπορεί να είναι περήφανοι γι' αυτό και εμείς για όλα αυτά τα επιτεύγματα του ρουμανικού λαού. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι και πάλι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν πολιτικές ελευθερίες και χρηστή διακυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εισακούονται όμως. Αντίθετα, το κυβέρνηση έχει οργανώσει πάταξη αυτών των ελευθεριών και των πολιτών και κατά της χρηστής διακυβέρνηση. Και τελικά ε, τίνει νομοθετικά να νομοποιήσει τη διαφθορά. Και μάλιστα ε, θα περισταλούν και οι διαμαρτυρίες. Θα πρέπει όμως μια προεδρία να δίνει το καλό παράδειγμα και να έχει και αξιοπιστία για να έχει ηγετική στάση. Έχετε ακόμα χρόνο να γίνετε το καλό παράδειγμα που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά ο χρόνος λιγοστεύει. Υπάρχουν πολλά ε, γεγονότα αυτό το εξάμεινο, το Brexit είτε έρθει είτε όχι, οι ευρωεκλογέ και ταυτόχρονα χρειάζεται και ένα όραμα μακροπρόθεσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά έχετε προγραμματίσει μια σύνοδο κορυφή το Μάιο, αλλά για να βοηθήσει αυτή η σύνοδο θα πρέπει να ασχολείται με τα φλέγοντα ζητήματα που θα πρέπει να λύσουμε. Τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή, πώ θα τη σταματήσουμε, πώ θα περάσουμε σε μια οικονομία χωρί διοξίδιο του άνθρακα, πώ θα έχουμε κοινωνικά δικαιώματα ε, που να είναι πραγματικό πραγματικότητα και όχι ωραία λόγια και πώς ε, θα ε, σταματήσουμε την υποχώρηση του κράτους δικαίου σε κάποια κράτη-μέλη. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ελπίζουμε να μας εκπλήξετε θετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Προεδρία της Ρουμανίας θα κληθεί να διαχειριστεί τη βαθιά οικονομική κρίση και τις τραγικές συνέπειες της τη διεύρυνση των ανισοτήτων τη συνεχή αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους και τη φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του κόσμου χωρίς να υπάρχει ελπίδα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η στατιστική για το 2017 ένας στους 7 συνταξιούχους είναι στο όριο της φτώχειας με αυξητική τάση. όλα αυτά όλα αυτά είναι που οδηγούν και τους λαούς στη μεγάλη αμφισβήτηση της ένωσης. δεν μπορεί λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση και η προεδρία σας να ζητούν την εμπιστοσύνη των λαών εν ώψη των ευρωεκλογών εάν δεν σταματήσει πρώτα η αιμονή στην πρόθεση των καταστροφικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών η στήριξη του συμφωνίου σταθερότητας η ευάθυνση της οικονομικής και δημοσιονομικής ένωσης καθώς και η λογική των προπολογισμών λιτότητας κυρία πρωθυπουργέ η gue ngl σας καλεί να αφουγκραστείτε τι ανησυχίε των λαών να προωθήσετε τι θέσει των προοδευτικών δυνάμεων του κοινοβουλίου για την ανάγκη ενίσχυση τη κοινωνική πολιτική. η κοινωνική ένδυα και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων που έγινε κανόνα, επιβάλλουν να επενδύσουμε άμεσα σε ένα κοινωνικό πυλώνα ο οποίο να έχει πραγματικό περιεχόμενο στη βάση των αναγκών τη κοινωνία. γιατί δυστυχώ σήμερα αποτελεί απλά συστηματικά ευχολόγια χωρίς καμιά δεσμευτική ισχύ. πρέπει επιτέλους να προηγηθούν μέτρα και να γίνουν επενδύσεις που να δώσουν όθηση στην πραγματική οικονομία να φέρουν ανάπτυξη προς όφελος των λαών και να ενισχύσουν την κοινωνική ε, συνοχή. αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να τεθούν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. ακόμα και η ψηφιοποίηση που τίθεται ως προτεραιότητα της προεδρίας σας πρέπει να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. εξίσου σημαντικό είναι να επιδειχθεί έμπρακτη αλληλεγγύη προ τα κράτη μέλη για μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση και όχι ενίσχυση τη λογική μια ευρώπη φρούριο. και τέλο αντί να δίνονται πακτολοί χρημάτων στην τουρκία και να τίθεται στην ημερήσια διάταξη αναβάθμιση τη τολωνιακή ένωση πρέπει να ασκηθούν πιέσει στην τουρκία να σταματήσει τι πειρατικέ ενέργειε σε βάρο τη κυριαρχία των κρατών μελών όπω είναι η ελλάδα και η κύπρος στο αιγαίο και στην ανατολική μεσόγειο. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και περισσότερα θέματα ε, με τα οποία ασχολείται. Έχουμε πολλές κοινέ αρχές και αξίες και τα συζητούμε ε, εδώ και καιρό. Τώρα έχουμε φτάσει στη φάση της εφαρμογής πολλών πολιτικών. Κυρία Πρωθυπουργέ, θα συμφωνούσατε ότι σήμερα, σήμερα το σημαντικότερο είναι να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ε, για ποιο λόγο ε, το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ονοποίηση έχει γίνει τώρα ενδιαφέρον για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τόσοι πολλοί Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και λοιποί να μην πάρουν τον ίδιο δρόμο. Κυρία Πρωθυπουργέ, για να απαντηθούν όλα αυτά τα ε, ερωτήματα. Δεν χρειάζονται και άλλα προγράμματα για οικονομική ανάπτυξη κλπ. Χρειάζεται να αλλάξει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ομάδα των ελευθεριών της άμεσης δημοκρατίας, ο κ. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα ε, μέχρι τώρα μου τράβηξαν την προσοχή. Πρώτον, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που έχει βάλει ε, θέμα τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων και συγχαρητήρια. Και μετά ο κύριος Μπούλμαν που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα ε, πέφτει στα παλιά πολιτικά πρότυπα και περνάει στην αντεπίθεση. Ε, αυτά είναι πράγματα παροχημένα, ανήκουν πια στην ιστορία. Τώρα αναλαμβάνεται την Προεδρία, παραδίδει η Αυστρία ε, είναι πολύ ε, μεγάλο και φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία διότι είναι δύσκολα τα θέματα και πραγματικά διαλέξατε θέματα καθόλου εύκολα, τα ακούσαμε προηγουμένως. Εγώ εκτιμώ πολύ τη Ρουμανία και τους Ρουμάνους. Έχω όμως κάποιες αμφιβολίες αν είναι σε θέση η κυβέρνησή σας να ε, δημιουργήσει και να διαμορφώσει μια λογική προεδρία και δεν ξέρω αν είστε αρκετά σταθερή κυβέρνηση, γιατί στην τρέχουσα θητεία είστε η τρίτη πρωθυπουργό. Ε, και δεν θα πρέπει να αναλωθούμε τώρα σε μάχες εξουσίας. Υπάρχει νομοθεσία ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς που προετοιμάζεται. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε όταν έρθει η ώρα και λήξει Προεδρία. Ο λόγος στον κύριο Ιβαν, Μην εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, σε αντίθεση με όσα σχολιάστηκαν και ακούστηκαν σήμερα, πιστεύω ότι αυτή η Προεδρία θα είναι μια Προεδρία επιτυχίας. Έχω την πεποίθηση ότι η Προεδρία της Ρουμανίας θα είναι μια επιτυχής Προεδρία, γιατί χρειαζόμαστε να πετύχει η Προεδρία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή. Πρέπει όλα όσα είπαμε και συζητάμε εδώ να λάβουν χώρα. Και γι' αυτό έχετε την υποστήριξή μου. Δεν ε, μας επιτρέπει ο χρόνος παρά να αναφέρουμε δύο θέματα τα οποία εγώ θεωρώ σημαντικά. Καταρχήν τα τρία τέταρτα των κρατών μελών αντιμετωπίζουν ε, όλο ένα και μεγαλύτερη σύγχρονη σκλαβιά στερούνται οι άνθρωποι την ελευθερία τους, εργάζονται χωρίς να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και πλήττεται όχι μόνο η Ρουμανία, αλλά στα τρία τέταρτα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντάμε αυτό το φαινόμενο. Μόνο στη Γερμανία είχαμε πάνω από 170.000 πολίτες που ήταν θύματα της σύγχρονης δουλείας. Το δεύτερο σημαντικό θέμα, μιλώνουμε για τη συνοχή. Σίγουρα χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους. Το άμεσο και το άμεσο κόστος της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει περίπου σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στη Ρουμανία ε, χάνουμε περίπου 40 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, πριν ήταν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ το κόστος στην Ιταλία 2 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται ετησίως. Στην Ισπανία 120 δις και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα ανακτήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνοχή για την οποία μιλάτε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στο θεματολόγιο της Προεδρίας. Καλησπέρα σε όλου. Προσκαλώ όλου του συναδέλφου να σέβονται το όριο του χρόνου, διότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Για Σούιτσα, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζω την εκπρόσωπο της Ρουμανικής ε, Κυβέρνησης. Χαίρομαι που αναλάβατε και την Προεδρία. Έχουμε την πρώτη Προεδρία του νέου